σωστή οικονομική προσέγγιση. Γι' αυτό υπάρχουν αυτά τα κονδύλια. Για να χρησιμοποιηθούν ε, τάχιστα για να ανταποκριθούμε σε μια κατάσταση κρίσης. Ευχαριστούμε. Κλείνει και αυτή η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου κατά τη μήνυ Ολομέλεια όπως σας είπα, τις πρώτες εβδομάδες του Μαΐου. Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα για τελευταίο της ημερήσιας διάταξης, που είναι η προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή για ειδικά μέτρα για, την, για τις γεωργικές αγορές. En, quien tiene la y vamos a iniciar el debate eh, Ας ε, δώσουμε το λόγο στον κύριο Στεφάν Λεφόλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι ήδη αργά. Και για να κλείσουμε, θα ήθελα καταρχήν να Ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του Παύλο που δεν μπορεί να παραστεί σήμερα γιατί όπως ξέρετε όπως και άλλοι δεν μπόρεσε να φύγει για να προσέλθει λόγω του ηφαιστείου. Το θέμα μας τίθεται από την κρίση που αντιμετωπίζει ο γεωργικός τομέας γενικότερα. Σήμερα ξέρουμε ότι υπάρχει κρίση και εκεί και ιδιαίτερα μείωση του αγροτικού εισοδήματος και των τιμών που πλήττει και τα δημητριακά και την κτηνοτροφία βόηο και χείριο κρέας και επίσης τους παραγωγούς ελαιολάδου όπως ο Πάολο Ντικάστρο καθώς και ιδιαίτερα τους γαλακτοπαραγωγούς. Και μπροστά σε αυτή την κρίση και τη μείωση των τιμών και εισοδημάτων είναι προφανές ότι η Επιτροπή Γεωργίας του Κοινοβουλίου θέλει να απευθυνθεί προς την Κομίσιον για να ζητήσει πληροφορίες ως προς το πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση αυτή και ιδιαίτερα τι μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν τους επόμενους μήνες για να βοηθήσουμε τους γεωργούς και ιδιαίτερα για να είναι λιγότερο πτυτικές, δηλαδή να αλλάζουν λιγότερο γρήγορα οι αγορές των γεωργικών προϊόντων. Τι φρονούν λοιπόν το Συμβούλιο και η Κομισιόν για την κρίση αυτήν και πώς σκοπεύουν να εφαρμόσουν τα ε, περίφημο γαλακτοκομικό ταμείο 300 εκατομμυρίων που έχει προβλεφθεί πώς θα χρησιμοποιηθεί. Όπως σας είπα, ολόκληρη η παραγωγή σήμερα, όλοι οι τομείς της γεωργίας πλήττονται από την κρίση. Άρα, τίθεται το ερώτημα ποια διευθέτηση μπορεί να γίνει των αγορών και πώς μπορεί να περιοριστεί αυτό, αυτή η μείωση των τιμών. Όταν ανεβαίνουν οι τιμές δεν παραπονείται κανείς, ιδίω η παραγωγή. Μόνο οι καταναλωτές και οι καταναλώτριες διαμαρτύρονται για την αύξηση των αγροτικών τιμών, γιατί έτσι περιορίζεται η αγοραστική τους δύναμη και ιδίως ως προς τα αγροτικά προϊόντα. Όταν όμως οι τιμές μειώνονται και μάλιστα σταθερά, η παραγωγή τότε ζημιώνονται, μειώνονται τα έσοδά τους και ιδιαίτερα μειώνεται η δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Γεωργίας να προετοιμάσει το μέλλον. Η γεωργία είναι βαριά βιομηχανία με μεγάλες επενδύσεις και κυρίως μακροχρόνιες. Πρέπει να σταθεροποιηθούν οι τιμές. Κύριε Επίτροπε, η Επιτροπή Γεωργίας και ο Πρόεδρος της Πάολο Ντικάστρο θέτουν δύο ερωτήματα. Πρώτον, ανακοινώσατε ορισμένα μέτρα πριν το τέλος του έτους για το γάλα. Μπορείτε να μας πείτε μερικά πράγματα επ' αυτού και πέρα από το γάλα τώρα. Πρέπει να ληφθούν και άλλα μέτρα και για άλλους τομείς. Και δεύτερο ερώτημα. Πώς θα μπορούσαμε μέσω πρόθεσμα να πούμε ότι η Κομισιόν θα προβλέπει, θα αποτρέπει τέτοιου είδους κρίσεις μείωσης των τιμών. Με ποιο μηχανισμό μπορεί κανείς να πει ότι θα περιορίζαμε και τις απότομες αυξήσεις και ιδιαίτερα τις βίαιες μειώσεις των τιμών. Τι προβλέπει να κάνει η Επιτροπή επ' αυτού. Τρία θέματα λοιπόν, τα γαλακτοκομικά και οι προοπτικές της και, και, οι, τους, και ιδιαίτερα πώς θα λυθεί αυτό το πρόβλημα της πτυτικότητας των τιμών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Λεφόλ. Ο Επίτροπος για να απαντήσει στα ερωτήματα αυτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ντικάστρο που εκπροσωπούσε ο κύριος Λεφόλ της Επιτροπής Γεώρ, Γεωργίας δηλαδή, Αγκρή. Πράγματι αναγνωρίζω ότι το εισόδημα των γεωργών έχει μειωθεί θεαματικά το 2009 και αυτό μετά και από προηγούμενη μίεση του 2008. Η κατάσταση αυτή λοιπόν είναι πρωτοφανής για την ευρωπαϊκή αγορά και εμφανίζεται μέσα σε πλαίσια ανοίγματο της ευρωπαϊκής αγοράς προς τη διεθνή και οφείλεται βέβαια και στην αδαρρύθμιση της ΚΑΠ. Η κατάσταση λοιπόν αυτή, η κρίση αυτή δεν αφορά μόνο τα γαλακτοκομικά. Πέρυσι είδαμε ότι αντιμετώπισαν ιδιαίτερες δυσκολίες η παραγωγή γαλακτοκομικών, αλλά ιδιαίτερα στις περιφέρειες όπου η παραγωγή σχεδόν περιορίζεται στα γαλακτοκομικά. Έτσι, η Κομισιόν πέρυσι έλαβε μέτρα πρώτον κινητοποιώντας μηχανισμούς που να σταματούσαν αυτή τη μείωση των τιμών ένα σημαντικό προϋπολογισμό 400, 400 εκατομμυρίων με παρεμβάσεις αλλά όπως το είπε και ο κύριος Λεφόλ δημιουργήθηκε και ένα γαλακτοκομικό ταμείο 300 εκατομμυρίων για να δώσει την ευκαιρία στα κράτη-μέλη να στηρίξουν τους ε, γαλακτοπαραγωγούς. Οι αποφάσεις αυτές λοιπόν λήφθησαν πέρυσι για να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη-μέλη να καθορίσουν κριτήρια με βάση τα οποία να κατανεμηθούν τα ποσά των ταμείων και να ωφεληθούν όσοι, θα, είχαν πληγεί περισσότερο. Τα καθόρισαν λοιπόν τα κράτη-μέλη αυτά τα κριτήρια και δεν χρειαζόταν έγκριση της Κομισιόν. Απλώς έπρεπε να πληροφορείται από τα κράτη-μέλη για τα κριτήρια που τα ίδια επέβαλαν. Όλα τα κράτη-μέλη από ό,τι ξέρω γνωστοποίησαν προς την Κομισιόν τι μέτρα θα ελάμβαναν με τι κριτήρια θα λαμβάνονταν τα μέτρα και θα κατανέμονταν τα ποσά του ταμείου και η κατανομή αυτή λοιπόν θα αρχίσει και θα συμπληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο. Μετά την πρώτη φάση δηλαδή την παρέμβαση στις αγορές για εξισορρόπηση της κατάστασης όπου νομίζω ότι φάνηκε ότι η παρέμβαση αυτή ήταν αποτελεσματική γιατί έγινε μια σχετική σταθεροποίηση των τιμών και οι διακυμάνσεις ε, δεν ήταν τεράστιες και μετά από την πρώτη εκείνη φάση χορηγείται τώρα αυτή η βοήθεια που σε λίγο θα πληρωθεί στους παραγωγούς. Αυτά είναι μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί τώρα. Επαναλαμβάνω όπως είπα και στην Επιτροπή Γεωργίας πρόσφατα ότι μετά από αυτά, αυτή την κατάσταση του περασμένου χρόνου συμπεράναμε ότι δεν θα περιμένουμε τη μεταρρύθμιση του 2013 της ΚΑΠ αλλά θα κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις για το γαλακτοκομικό τομέα Βάσει των συμπερασμάτων της ομάδας υψηλού επίπεδου που ακόμη δεν τελείωσε τις εργασίες της που δημιουργήθηκε πέρυσι για να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση. Η ομάδα υψηλού επίπεδου λοιπόν θα υποβάλει τον Ιούνιο τα συμπεράσματά της και αμέσως μετά τον Ιούλιο θα προτείνω συζήτηση μεταξύ Υπουργών Γεωργίας και Επιτροπής Γεωργίας στο Κοινοβούλιο και σε αυτή τη βάση Μέχρι το φθινόπωρο και το τέλος του έτους θα υποβάλω προτάσεις που θα μας επιτρέψουν ειδικά για το γαλακτοκομικό τομέα όπου υπήρξε η δυσκολότερη κατάσταση που θα μας επιτρέψουν πως στο μέλλον να αποφεύγονται στο εξή τέτοιου είδους κρίσεις και άρα θα προτείνω λύσεις όχι απλώς βραχυπρόθεσμες αλλά και μέσω μακροπρόθεσμες και αυτά τα μαθήματα θα τα εφαρμόσουμε και για άλλους αγροτικούς τομείς όπου χρειάζεται παρέμβαση. Θα σας δώσω περισσότερα στοιχεία γιατί η Κομισιόν παρακολουθεί όλους τους αγροτικούς τομείς και με βάση τα στοιχεία που έχουμε για τις παρεμβάσεις και τους μηχανισμούς που διαθέτουμε θα προσπαθήσουμε να αποφεύγονται τέτοιες καταστάσεις στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Θα το προσέξω ιδιαίτερα και θα επανέλθω αργότερα. Ευχαριστούμε και σας καλωσορίζουμε στην νυχτερινή μας ολομέλεια. Αρχίζουμε με τον γύρο των ομιλητών εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Γιάρ, εξ ονόματος του ΕΛΚ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε και κύριοι. Θεωρώ ότι η κατεύθυνση της Γεωργίας προς μία προς ένα προσανατολισμό της ε, οικονομίας της αγοράς είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει την ευρωπαϊκή γεωργία. Τα πρώτα στοιχεία αυτής της πολιτικής τα είδαμε από φέτος τον Ιανουάριο. Μεγαλύτερη σταθερότητα τιμών, καλύτερα εισοδήματα για τους αγρότες, Παρόλα αυτά είχαμε και κάποιες μεγάλες διακυμάνσεις τιμών και μείωση του εισοδήματος των γεωργών. Δυστυχώ στο μέλλον θα πρέπει να αντιμετωπίζουν αυτή τη μεταβλητότητα των τιμών οι αγρότες σε όλους τους τομείς, όχι μόνο των γαλακτοκομικών. Και η αντιμετώπιση που πρέπει να έχουμε εμείς δεν πρέπει να είναι γραφειοκρατική. Μας ενδιαφέρουν λοιπόν πιθανές παρεμβάσεις ε, όπως ε, ενισχύσεις εξαγωγής ε, οι οποίες ενδεχομένως να χρησιμοποιούνται μόνο σε περιστάσεις εκτάκτου ανάγκης και υποφυσιολογικές συνθήκες να είναι στο μηδέν. Απλά πρέπει να υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες και να είναι έτοιμες να τις χρησιμοποιήσουμε όπου απαιτείται. Είναι σημαντικό να έχουμε μία ισοτιμία στην αγορά για τους γεωργούς, για τη γεωργία. Αναφερθήκατε στις οργανώσεις των παραγωγών. Θεωρούμε ότι οι οργανώσεις παραγωγών χρειάζονται ένα καλύτερο νομικό πλαίσιο και την δυνατότητα να λαμβάνονται μέτρα προκειμένου να μην έχουμε μόνιμες συνέπειες για τους καταναλωτές. Ευχαριστώ κύριε Σταραμπέλα, δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για τα πρώτα σας βήματα ως Επιτρόπου Γεωργίας. Σας ακούσαμε στην Επιτροπή μας, ακούσαμε τις ελπίδες σας και όντως θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν εχθρούς οι Γεωργοί μας και δεν βλέπουν προοπτικές καθώς ε, οι επενδύσεις ε, για τους ε, πιο νέους υπολογίζονται πλέον με χρονικό ορίζοντα 20-30 ετών. Αυτή τη στιγμή εδώ και έξι μήνες μαζί με τον συνάδελφο Λεφόλ είχαμε υπογράψει μια τροπολογία για το γάλα για μείωση στο 1%. Αυτό όμως ουσιαστικά τελικά καταρρίφθηκε, απορρίφθηκε με περίπου 250 ψήφους κατά. Σήμερα έχουμε συνεδρίαση της ομάδας υψηλού επίπεδου, αλλά τελικά αυτό που ακούω είναι ότι ναι μεν εκπροσωπούνται πολλά σημαντικά άτομα και μεταξύ των οποίων διανομής και παραγωγή, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και μία άλλη σημαντική ομάδα, τους μεταποιητές, γιατί αυτοί είναι που έχουν τα μεγαλύτερα κέρδη, μεγαλύτερα και από τους διανομής. Δεν πρέπει λοιπόν να τους ξεχνάμε σε αυτή τη συζήτηση. Πέρα και από τον ε, τομέα του γάλακτος βλέπουμε ότι η μεταβλητότητα των τιμών φορά όλους τους τομείς και είναι αλήθεια ότι αυξάνονται πολύ οι τιμές. Δεν είναι πάντα καλό για τους παραγωγούς γιατί οι καταναλωτές επιλέγουν υποκατάστατα προϊόντα και όταν πέσουν οι τιμές ενδεχομένως δεν επανέρχονται στα αρχικά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν χρειαζόμαστε μέτρα, μέτρα ρυθμιστικά που τα αναμένουν με ανυπομονησία η παραγωγή. δώσω τον Πρασίνων για μισή λεπτά. Ο κύριος Χόισλινγκ έχει το λόγο. Κύριε Επίτροπε, πρόσφατα Βλέπουμε, άμα πάμε στην Ήπεθρο, ότι η γεωργοί είναι πάρα πολύ απογοητευμένοι και δεν μπορούμε να αναμένουμε το 2013 για να εξεύρουμε λύσεις. Θα πρέπει να τις βρούμε τώρα, διότι οι διαμαρτυρίες θα φτάσουν πολύ γρήγορα στις Βρυξέλλες. Θα έρθουν οι γεωργοί στις Βρυξέλλες αν χρειαστεί στον τομέα των γαλακτοκομικών ε, θεώρησα ότι οι απαντήσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων ήταν μια απάντηση αλλά ίσως όχι κατάλληλη για την κρίση στον τομέα των γαλακτοκομικών. Είπαμε να απομακρυνθούμε από μια λύση κανονισμού. Και βεβαίως οι αγρότες δεν προσγειώθηκαν στα μαλακά μετά από αυτό. Θα πρέπει να δούμε τι μέτρα μπορούμε να λάβουμε εμείς ως πολιτικοί έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να ξαναμπούν στο παιχνίδι και οι αγορές να λειτουργούν κανονικά. Κάτι το οποίο δεν γίνεται μετά την κρίση των γαλακτοκομικών. Θα πρέπει να βρούμε απαντήσεις. Γίνονται πολλές συγχωνεύσεις στον τομέα των γαλακτοκομικών και βλέπω ότι στη Νότια Αγγλία, για παράδειγμα, έχουμε ζωικά κεφάλαια ε, της τάξης των 8.000 κεφαλών, ενώ ε, οι μικρότερες περιφέρειες δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Δεν υπάρχουν ίσοι όροι ε, παιχνιδιού. Κινούμεθα προς τα πρότυπα των ΙΠΑ, δηλαδή των μεγάλων εκμεταλλεύσεων θα πρέπει να αναγνωρίσουμε αυτή την τάση. Συμφωνώ με τον κύριο Γιάρ επί ενός θέματος. Χρειαζόμαστε ένα νομικό πλαίσιο, σαφές νομικό πλαίσιο για τους γεωργούς, διότι είναι ο πιο αδύναμος κρίκος στην εμπορική αλυσίδα. Διαφορετικά θα πρέπει να υποστούμε το ντάμπινγκ των τιμών και θα πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε για τους γεωργούς μας και να οργανώσουμε τις αγορές κατά καλύτερο τρόπο για να μην πλήττονται οι μικρές επιχειρήσεις. Θα πρέπει να δούμε πώς γίνονται τα πράγματα αλλού. Πρέπει να ρυθμίσουμε τις αγορές μας. Προχωρήσαμε πολύ μακριά με την απορρίθμιση τα πρόσφατα χρόνια και η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να δει πού γίνονται τα πράγματα διαφορετικά και γιατί. Γιατί το καναδικό μοντέλο ίσως θα ήταν το καλύτερο. Δεν λέω ότι πρέπει να τους αντιγράψουμε τους Καναδούς, αλλά να δούμε πώς λειτουργεί το δικό του σύστημα. Αυτό αφορά και τις περιφερειακές αγορές. Δεν θα πρέπει να βασιστούμε στο 5% των προϊόντων που αγοράζονται και πολλούνται στις ε, παγκόσμιες αγορές. Ως προς τις εξαγωγές και τις τιμές παρέμβασης δεν θα πρέπει να είναι καθημερινά μέτρα. Κλείνουμε αυτό το γύρο με τον κύριο Νίκολσον εξ ονόματος των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να πω καταρχάς ότι χαίρομαι που μπορούμε να έχουμε σήμερα τη συζήτηση αυτή. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα έγκαιρη. Τώρα που η οικονομική κρίση δημιούργησε τρομερά προβλήματα σε πολλούς γεωργούς και η μεταβλητότητα έδειξαν ότι μπορεί να δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στις αγορές. Η μεταβλητότητα των τιμών είναι κάτι που εμφανίζεται πλέον αρκετά συχνά και δεν έχει πάντα να κάνει με παράγοντες που εξαρτώνται από εμά. Για παράδειγμα, άνοδος τιμών των πετρελαίου και παγκοσμιοποίηση. Εμείς όμως πρέπει να μπορέσουμε να αντιδράσουμε γρήγορα. Ένα σύστημα διαχείρισης και στήριξης των αγορών που θα μπορούσε να μειώσει τις ε, επιπτώσεις είναι απαραίτητη και διαφορετικά θα δούμε και άλλους ε, γεωργούς να φεύγουν από τη γεωργία και να βλέπουν το εισόδημά τους να καταρρέει. Θεωρούμε ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι Πρώτον, να έχουμε ένα ελάχιστο δίκτυ ασφαλείας για όλους τους τομείς που είναι ευαίσθητοι στις μεταβολές των τιμών. Δεύτερον, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ό,τι εργαλεία και αν χρησιμοποιήσουμε θα πρέπει να μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε άμεσα και αποτελεσματικά οποτεδήποτε υπάρχει κρίση. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλές συζητήσεις για το ότι χρειάζονται δίκαιο εισόδημα οι γεωργοί μας για την παραγωγή τους. Αυτό το θέμα αφορά και τους παραγωγούς και τους καταναλωτές. Εφόσον θα έχουμε σύντομα μεταρρύθμιση της γεωργικής πολιτικής θα μπορέσουμε να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Βεβαίως δεν πρέπει να μειώσουμε και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας. Ωστόσο η μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής θα πρέπει να μας δώσει την δυνατότητα να αντιμετωπίζουμε τις κρίσεις και να σταθεροποιούμε τις αγορές αλλά και να δίνουμε δίκιο εισόδημα στους αγρότες μας. Ο πρώτος ομιλητής για δύο λεπτά είναι ο συνάδελφος ο κύριος Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκκινώ από την παραδοχή ότι παρατηρείται μεγάλη αστάθεια στι γεωργικέ αγορέ και σημαντική πτώση των τιμών βασικών γεωργικών προϊόντων. Παράλληλα, σημειώνεται αύξηση των τιμών καταναλωτή και ουσιώδη ε, μείωση του αγροτικού εισοδήματο. Κατά τη γνώμη μου, η ΚΑΠ, συνεπία των αναθεωρήσεων και με την αποσύνδεση των ενισχύσεων, είναι αρκούντο προσανατολισμένη στην αγορά η μείζον πρότασή μου και θέλω να την καταστήσω σαφή είναι ότι ο γεωργικός τομέας δεν μπορεί να αφαιθεί πλήρως στους κανόνες της αγοράς. παράγει δημόσια αγαθά απαιτείται δημόσια ευρωπαϊκή χρηματοδοτική στήριξη. και δεν μπορώ να παρακολουθήσω την αντίφαση της επιχειρηματολογία συναδέλφων οι οποίοι εδώ προτάσουν τον προσανατολισμό στην αγορά αλλά στις χώρες τους συντηρούν καλλιεργούν επιτείνουν έναν καταναλωτικό εθνοκεντρισμό έναν καταναλωτικό πατριωτισμό. ωστόσο τα ισχύοντα μέτρα ασφαλείας μέτρα διαχείρισης αγοράς μάλλον δεν παρέχουν το απαραίτητο δίκτυο ασφαλείας το είπε αυτό και ο προλαλής σας συνάδελφος ο κύριος Νίκολσον. Χρειαζόμαστε συμπληρωματικά μέτρα περισσότερο ευέλικτα και αποτελεσματικά. Μέτρα τα οποία θα αγγιώνται σε περιόδους κρίσεων τη σταθερότητα των αγορών επίσης κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να εξοπλίσουμε την καπ με έναν δημοσιονομικό μηχανισμό για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσεων αν θέλετε ένα ταμείο διαχείρισης ε, κρίσεων. η εγγύηση του εισοδήματος των ε, παραγωγών προϋποθέτει πέραν των άλλων και τη διασφάλιση της διαφάνειας στην εφοδιαστική ε, τροφική αλυσίδα και δεν μπορούμε και τελειώνω να περιοριστούμε στο σχεδιασμό μελλοντικών εργαλείων αγοράς μετά το. 2013. Γνωρίζουμε ότι η κατάσταση πέραν του τομέα του γάλακτος είναι κρίσιμη και σε άλλους τομείς ιδιαίτερα σημαντικούς οι οποίοι διαφοροποιούνται από γεωγραφική περιοχή σε γεωγραφική περιοχή εντός της Ευρώπης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριο Ταμπάζδη για δύο λεπτά. Κύριε Σόλος, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι έχουμε να κάνουμε με μία πολύ προβληματική συλλογιστική. Ο κύριος Ταραμπέλα και άλλοι μίλησαν για το γεγονός ότι το θέμα αυτό σχετίζεται με την διατροφική αλυσίδα που απασχολεί και την έκθεση Μποβέ. Και πώς μπορούμε να εγγυηθούμε μια δίκαιη κατανομή μεταξύ, κατανομή μεταξύ παραγωγών και διανομέων, καθώς και μεταποιητών. Θα πρέπει να βρούμε μια μακροχρόνια λύση η μία δυνατότητα αναφέρθηκε από τον κύριο Γιάρ. Να δούμε δηλαδή, να βασιστούμε στη νεοφιλελεύθερη τάση που προσπάθησε να αποδομήσει το σύστημα παρέμβασης. Θα πρέπει να μας απασχολήσει αυτό το σύστημα παρέμβασης και η γαλλική πρόταση βασιζόταν στο, στην, στο αντικυκλικό ρυθμιστικό πλαίσιο, αλλά είπα, είναι τόσο μεταβλητή η αγορά που θα πρέπει να δούμε όλες τις δυνατότητες. Τρίτον, η χρηματιστηριακή προσέγγιση. Έγινε μία τηλεδιάσκεψη με σύστημα online με το χρηματιστήριο για να δούμε κατά πόσο τα χρηματιστήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτό το τομέα. Και θα ήθελα να πω στον Επίτροπο Τσόλος ότι στις βαλτικές χώρες δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Μετά η Γαλλική Προεδρία μίλησε για ένα ευρωπαϊκό σύστημα ελέγχου των τιμών, παρατήρησης των τιμών. μπορούμε να εφαρμόσουμε το θέμα μεταρρύθμισης των οποροκυπευτικών έτσι ώστε σε περίπτωση κρίσης να εφαρμοστεί αυτό το σύστημα με βάση τα ταμεία και θα χρησιμοποιηθούν πολλά ποσά. Θα πρέπει να δούμε όλες τις δυνατότητες, διότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να ρυθμίσει τις αγορές. Ο κύριος Βοζικόφσκι δεν είναι παρόν. Ο Μισελ Νταντέν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, γνωρίζετε πολύ καλά ότι η γεωργία είναι ένας οικονομικός τομέας με ιδιαιτερότητες και γι' αυτό ορισμένες φορές είναι απαραίτητη η δημόσια παρέμβαση ή τουλάχιστον επιθυμητή από τους παραγωγούς, τους καταναλωτές και τους πολίτες. Και αυτό δικαιολογείται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκοσμίω για τρεις λόγους. Καταρχάς γιατί τα γεωργικά αγαθά αλλά και οι αγορές είναι ασταθή. Επίσης δημιουργούνται και μη εμπορεύσιμα αγαθά, όπως για παράδειγμα η κοινωνική σταθερότητα στην Ήπεθρο και η απασχόληση. Επίσης έχουμε ποικιλόμορφες συνέπειες της γεωργίας. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε εμείς. Γνωρίζετε ότι θα σας δώσω κάποια στοιχεία μάλλον για τον τομέα της κτηνοτροφίας. 800 από τις επιχειρήσεις ενός μήνατος της Γαλλίας έχει υπερχρέωση ορισμένες φορές πάνω από το 100%. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή έχουμε αποκεφαλισμό της γεωργίας και άρα έχουμε ένα εκρηκτικό κοκτέιλ εξαιτίας της μείωσης των ενισχύσεων και της αύξησης των περιορισμών. Σίγουρα πρέπει να γίνουν αλλαγές. Όμως θα ήθελα να τονίσω κάποιες ε, αποφάσεις της Επιτροπής και των συναδέλφων σας κύριε Επίτροπε που οδηγούν στο γεγονός ότι παρά την κατάσταση της αγοράς βλέπουμε προβλήματα για όλους τους τομείς, κρέατος, λαχανικών κτλ. Και βλέπουμε να θυσιάζονται και η παραγωγή των ε, άκρως απόκεντρων περιοχών για χάρη των, της Λατινικής Αμερικής. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σιλβέστρης, δύο λεπτά. Προέρχομαι από τη Νότια Ιταλία και η περιφέρειά μας βασίζεται στις μεσογειακές, ε, στη μεσογειακή παραγωγή. Οποροκυπευτικά, ελαιόλαδο, αλλά έχουμε και πολύ μεγάλο ζωικό κεφάλαιο. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις μεσογειακές καλλιέργειες. Στις περιφέρειες μας βλέπουμε την απερίμωση των εκμεταλλεύσεων. Υπάρχει εγκατάλειψη των εκμεταλλεύσεων λόγω απερίμωσης. Δηλαδή βλέπουμε παράσιτα εκεί όπου υπήρχαν οπορώνες. Το 1995 η ελαιοπαραγωγή λάμβανε 170.000 λίρες, δηλαδή 30 ε, ευρώ τα 5 κιλά. Τώρα βλέπουμε ότι το ελαιόλαδο στοιχίζει 2 ευρώ το λίτρο. Άρα δεν μπορεί να καλυφθεί ούτε το κόστος. Είναι υπερχρεωμένες οι γεωργικές επιχειρήσεις. Και το ελαιόλαδο στη λιανική το βλέπουμε 2 ευρώ ή και κάτω, ενώ χονδρική το αγοράζουμε 2 ευρώ και πάνω. Θα ήθελα ο κανονισμός 2568 κάθετος 91 να αλλάξει, γιατί ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πλήττονται οι παραγωγοί. Δεν μπορούμε να εθνικοποιήσουμε τις επιδοτήσεις στην προσεχή ΚΑΠ, διότι χωρίς άμεσες επιδοτήσεις η μεσογειακή μας γεωργία θα καταπέσει. Όποιος σήμερα έχει μία έκταση δεν την κέρδισε στο λότο την ε, έχει επειδή την έλαβε από τον ε, πατέρα του, από τους γονείς του. Έχει φτύσει αίμα και δεν μπορεί να τελειώσει τη ζωή του υπερχρεωμένος. Θα πρέπει να βοηθήσουμε την ε, γεωργία μας. Ένα ζητάει το λόγο μας στα πλαίσια του Catch the Eye. Οι άλλοι θα κοιμηθούν ή κοιμούνται. Έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η σταθεροποίηση των αγορών πρέπει να είναι ένας από τους βασικούς στόχους της κοινής πολιτικής. Νομίζω ότι οι περισσότεροι συμφωνούμε. Επίσης χρειαζόμαστε μέτρα για την αγορά αλλά και μέτρα ασφαλείας για τους παραγωγούς καθώς και για όλους τους κρίκους της αλυσίδας. Από ό,τι φαίνεται από το 2014 και μετά τα πράγματα θα γίνουν ακόμη πιο προβληματικά με αύξηση των εισαγωγών από τρίτες χώρες. Ο Επίτροπος μας είπε ότι θα ληφθούν μέτρα ήδη πριν το 2013. Οπότε τώρα πρέπει να εξετάσουμε το πώς θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα νέα μέτρα για την αγορά και να βοηθήσουμε τις οργανώσεις αλλά και να αυξήσουμε τη διαφάνεια στην αγορά. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Θέλετε να παρέμβετε μέσα στα πλαίσια της παρέμβασης ενός λεπτού ή γιατί σηκώσατε την ε, καρτέλα σας. Ωραία, έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, έχω μία μελέτη εδώ ενός γερμανικού γεωργικού φορέα και βλέπουμε μία μελέτη μεγάλης εμβέλειας που έχουν δευτερογενή δραστηριότητα στις γεωργικές επιχειρήσεις το 2008 9 η κατάσταση έχει επιδεινωθεί για αυτές τις επιχειρήσεις τις 18.000 γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οικογενειακές επιχειρήσεις από 45.000 έπεσε το εισόδημα στις 34.000, δηλαδή έπεσε κατά, 30, κατά 24%. Και ιδιαίτερα επλήγει ο γαλακτοκομικός τομέας. Άρα τα εισοδήματα έπεσαν μεταξύ 20 και 30% για αυτές τις επιχειρήσεις. Ο πρόεδρος διακόπτη και δίνουμε το λόγο στον Επίτροπο, στον κύριο Τσόλος. Για να παρέμβει με βάση τις προγενέστερες ομιλίες. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ ότι η συζήτηση που μόλις άκουσα μας αποδεικνύει πως η κρίση στον τομέα του γάλακτος μπορεί να μας οδηγήσει σε διδάγματα όπως είπε και ο κύριος Λεφόλ στην αρχική του παρέμβαση, προκειμένου να καταλήξουμε σε μηχανισμούς ρύθμισης της αγοράς για την κοινή γεωργική πολιτική μετά το 2013. Εγώ θεωρώ ότι η κοινή γεωργική πολιτική, λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία της γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα κοινά στοιχεία και να προτείνει μέτρα που θα μας επιτρέψουν να επιτύχουμε τους στόχους της κοινή γεωργικής πολιτικής, δηλαδή σταθερότητα του εισοδήματος και χωρίς προβλήματα τροφοδοσία της αγοράς. Αυτή είναι η στόχη της συνθήκης της Λισαβόνας και πρέπει να τους επιτύχουμε μαζί με τους υπόλοιπους. όσον αφορά τα μέτρα ρύθμισης της αγοράς που θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν να παρεμβαίνουμε σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη μεταβλητότητα των τιμών και την αστάθεια των αγορών. Θα υπάρξουν προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κοινή γεωργική πολιτική μετά το 2013. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ήδη εργαζόμαστε επί του θέματος και ότι συνειδητοποιούμε ότι πέρα από τις άμεσες ενισχύσεις που πρέπει να διατηρηθούν με συγκεκριμένα κριτήρια χρειάζονται και μηχανισμοί διαχείρισης της αγοράς που μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο. Βεβαίως πρέπει να αφήσουμε και τις αγορές να λειτουργούν όποτε μπορούν να λειτουργούν. Όμως συμφωνώ και με όσους είπαν ότι οι ιδιαιτερότητες του τομέα της ε, γεωργίας δικαιολογούν κάποιες ε, παρεμβάσεις του δημοσίου προκειμένου να υπάρξει καλύτερη λειτουργία αλλά όχι όταν λειτουργεί σωστά η αγορά. Στα πλαίσια λοιπόν της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής του μετά το 2013 θα εξετάσουμε αυτά τα θέματα. Γνωρίζω ότι πέρα από τον τομέα του γάλακτος υπάρχουν και άλλοι τομείς που υποφέρουν ιδιαίτερα. Για παράδειγμα ο τομέας των οπαραχαλεχανικών που αντιμετώπισε μεγάλη αστάθεια τιμών. Υπήρξε μεταρρύθμιση του τομέα των οπαραχαλεχανικών ε, στο πρόσφατο παρελθόν και τώρα αξιολογούμε τα αποτελέσματα που έχουν να κάνουν μεταξύ άλλων και με τις συνέπειες ε, στις οργανώσεις των παραγωγών αλλά πρέπει να δούμε και τις συνέπειες για τους καταναλωτές. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να επιτρέψουμε στους παραγωγούς να κάνουν καλύτερες διαπραγματεύσεις για τις τιμές, για τα συμβόλαιά τους, προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη σταθερότητα της προμήθεια στην αγορά με ιδιωτικές συμβάσεις. Επαναλαμβάνω, πρέπει να επιτρέψουμε στην αγορά να λειτουργήσει όποτε αυτό είναι δυνατό, αλλά παράλληλα να δώσουμε τη δυνατότητα στο δημόσιο τομέα να επεμβαίνει όπου χρειάζεται. Γιατί δεν μας ενδιαφέρει μόνο να έχουν προϊόντα οι αγορές αλλά να μπορούμε να προσφέρουμε και ένα δημόσιο αγαθό. Και στα πλαίσια αυτού του στόχου μπορεί να χρειαστεί και βοήθεια. Για τα ερωτήματα που έχουν να κάνουν με τη διατροφική αλυσίδα τώρα. Η δυνατότητα διαπραγμάτευσης για καλύτερη κατανομή της προστιθέμενης αξίας και εκεί έχει ασχοληθεί με το θέμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενώ συνεχίζονται οι συζητήσεις και στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο οπότε με βάση όλα αυτά θα μπορέσουμε να καταλήξουμε πιστεύω σε προτάσεις που θα μας επιτρέψουν να βρούμε τους μηχανισμούς που θα δώσουν τη δυνατότητα στους παραγωγούς να διαπραγματεύονται καλύτερα τα περιθώρια κέρδους τους. Νομίζω ότι απάντησα σε όλα τα ερωτήματα σε όλα τα προβλήματα που με επισημένθηκαν. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι που μου δώσατε τη δυνατότητα να σας απευθύνω το λόγο. Είναι σημαντικό να υπάρξει δημόσιος διάλογος πριν περάσουμε στη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής για την περίοδο μετά το 2013 και πιστεύω ότι μετά από αυτό το δημόσιο διάλογο και μετά τις εργασίες και του Κοινοβουλίου θα επανέλθουμε με ανακοίνωση της Επιτροπής το φθινόπωρο χώρο για τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής και θα πρόκειται για μια πρόταση που θα δίνει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους ε, παραγωγούς για το σύστημα. Ευχαριστώ πολύ. Κλείνουμε τη συζήτηση καθώς και τη σημερινή Ολομέλεια. Η επόμενη θα λάβει χώρα αύριο 21 Απριλίου Ξέρετε, από τις 9